Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, please take your seats. We will start voting in one minute. Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Πρώτη είναι η έκθεση Γκάμπριελ. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία.